Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη ακολουθεί η εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω λάβει τις εξή υποψηφιότητες, τις οποίες τώρα θα διαβάσω. Με αλφαβητική σειρά. Έχουν υποβληθεί οι υποψηφιότητες των... Ρομπέρτα Ντουρόν, Καράς miguel angel martinez martinez edward mcmillan scott georgios papastamkos gianni pittella ani podimata jacek protasiewicz laszlo surjn indrek tarand alejo vidal quadras oldrich vlasak und rainer Οι υποψήφιες και οι υποψήφοι μου είπαν πως προτείνονται βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη τους. Παρακαλώ καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι γιατί θα περάσουμε στην διεξαγωγή της ψηφοφορία. Όσου, όσους ενοχλώ παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα. Κύριε Ντόλ. Κύριε Ντόλ. Εάν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ καθίστε. Καλό θα ήταν, νομίζω, είστε και να δώσετε και το καλό παράδειγμα ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην ψηφοφορία. Wahlhelfer bei diesem Wahlgang sind dieselben wie bei der Wahl des Präsidenten. Ich ersuche die. Οι ψηφολέκτε είναι οι ίδιοι με την ψηφοφορία του Προέδρου. Παρακαλώ λοιπόν να προσέλθουν κοντά στην κάλπη και θα ψηφίσουν τελευταίοι. είναι όλοι οι συνάδελφοι στην αίθουσα. Είναι η Μπορσελίνο Ζόγκορ, Παπαναγιώτοφ, Ποκ, Μπάγκο, ο κύριος Καλινόφσκι, ο κύριος Κάλβιν και ο κύριος Περέγιο Ροντρίκες. Παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις σας. Απουσιάζει κάποιος από αυτούς που ανέφερα βεβαίως. Ναι, περίεργη ερώτηση, δεν μπορεί να απαντήσει ο ίδιος. Ξέρετε αν αποσιάζει κάποιο από αυτού που ανέφερα. Δεν ξέρω. Δεν είναι μυστική διαδικασία. Παρακαλώ, λάβετε θέση κοντά στις κάλπες, αλλιώς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ε,

Μπορσελίνο είναι εδώ. Κυρία Μπορσελίνο είναι εκεί, εκεί πάνω. Go. Ja? Okay, der mir. Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind alle Wahlhelfer? Είναι όλοι λοιπόν στι θέσει του. Μάλλον ναι. Ο αριθμός τώρα των υποψηφίων ξεπερνάει τον αριθμό των θέσεων αντιπρόεδρων. Οπότε, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, πρέπει να ψηφίσουμε σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Γι' αυτό θα ξαναδιαβάσω το άρθρο 15 παράγραφος 1. Μετά την εκλογή των, ε, του Προέδρου εκλέγονται οι αντιπρόεδροι με ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία στον αριθμό των 14 και κατά τη σειρά των ψηφων ο αριθμό των εκλεγένων αντιπρόεδρων. Και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν, ε, που έχουν ε, συγκεντρώσει κτλ. Αν ο αριθμό των εκλεγέντων είναι μικρότερο από τον αριθμό των ε, πλήρωση εδρών, διεξάγεται και δεύτερη ψηφοφορία κτλ. Εάν δεν ε, πληρωθούν και οι 14 θέσεις με το πάνω από το ίμιση των ε, έγκυρων ψήφων, λαμβάνει χώρα δεύτερη ψηφοφορία. Και εξακολουθεί να απαιτείται η πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων για να εκλεγεί κανείς. Εάν και τότε δεν συγκεντρώσουν 14 την απαραίτητη πλειοψηφία, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία στην οποία ισχύει η σχετική και όχι ε, απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφία εκλεγέντες θεωρούνται οι πρεσβύτεροι από τους υποψηφίους. Μπορείτε λοιπόν να σταυρώσετε 14 υποψηφίους. Παρακαλώ να το κάνετε αυτό στα προτυπωμένα κουτάκια δίπλα στο κάθε όνομα, αλλιώς τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα. Μπορείτε λοιπόν να σταυρώσετε μέχρι 14. Εάν σταυρώσετε 15 είναι άκυρο. Βεβαίως αν θέλετε μπορείτε να σταυρώσετε μόνο έναν ή μία. Το πολύ λοιπόν 14. Εάν κάνετε λάθος Εάν αλλάξετε άποψη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πετάτε το ψηφοδέλτιο, ζητάτε ένα καινούριο ψηφοδέλτιο. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείτε να διορθώσετε το λάθος. Τυπλώστε λοιπόν το ψηφοδέλτιο, βάλτε το σφάκελο και ρίχτε το στην κάλπη. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τη διαδικασία πλην του συναδέλφου Κονπεντίτ. Όχι. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν τώρα τους κλητήρες να μοιράσουν τα ψηφοδέλτια. Συμπληρώστε τα και κατευθυνθείτε προς τις κάλπες. Ευχαριστώ πολύ.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 Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Ψήφισαν και οι ψηφολέκτες. Από ό,τι βλέπω, ναι. Άρα φτάσαμε στο πέρας της ε, ψηφοφορίας. Παρακαλώ λοιπόν να περάσουν οι ψηφολέκτες για την καταμέτρηση στην αίθουσα R01101. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι την ώρα την οποία θα δείτε στις οθόνες.